Euh, θα αρχίσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας και σας ζητώ ε, να δεχτείτε την ε, συγνώμη του πρέσβος ε, κυρίου Χάμπερ, ο οποίος θα έπρεπε να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ο κύριος Χάμπερ είναι άρρωστος, όπως και πολύ μεταξύ μόνο, ο πρόεδρος ας πούμε ε, δεν ε, αισθάνεται και πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας, μας ζητά ο κύριος Χάμπερ να τον συγχωρήσουμε. Είναι διοικητής πολιτικών δράσεων της ΕΠΣΣ και δεν θα είναι εδώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις υπόλοιπες ε, συνεδρίες, τα υπόλοιπα θέματα μας. Ε, και μια και δεν θα έχουμε το θέμα των μη στρατιωτικών αποστολών και μια και έχουμε και την Άννα μεταξύ μας, ε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια σχετικά με την αποστολή που κάναμε 15 μέρες πριν στη Λιβύη. Έγινε αποστολή λοιπόν ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, στην Βενγάζη και στην Τρίπολη πριν από δύο εβδομάδες. Ήταν η Άννα ως εισηγήτρια για τη Λιβύη, εγώ ο ίδιος ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας, ο πρόεδρος Σαλαφράνκα που προείδρευε ο κύριος Παντζέρη επίσης, ε, είμαστε πέντε ε, στην Τρίπολη και στην ε, Βενγάζη έτσι ώστε να κάνουμε μια αποστολή, είχαμε μια αποστολή πάρα πολύ πυκνή, πολλές επισκέψεις, επισκεφθήκαμε, συζητήσαμε πάρα πολύ κόσμο μεταξύ των οποίων ε, τον ίδιο τον πρόεδρο του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, συναντήσαμε επίσης ε, πολλούς εκπροσώπους ε, της κοινωνίας των πολιτών, τον Γιάν Μάρτιν, συντονιστή του ΟΗΕ, καθώς επίσης και άλλους εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών. Ε, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είχαμε πάρα πολλές συναντήσει. Ε, μετά το πέρας της αποστολής μας στείλαμε ε, επιστολή εις ε, την υπεύθυνη της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι ότι θα έχετε όλοι λάβει ένα αντίγραφο της επιστολής αυτής. Στην επιστολή αυτή λοιπόν αναφερθήκαμε κυρίως στα θέματα ασφάλειας γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν περισσότερο πρέπει να πω ότι η πρώτη διαπίστωση όσον αφορά την κατάσταση στην ε, Λιβύη, ε, η πρώτη διαπίστωση λοιπόν είναι λιγότερο καταστροφική αν θέλετε, ε, από ό,τι διαβάζουμε ή βλέπουμε σε πολλά μέσα ενημέρωσης που τίνουν να παρουσιάσουν την κατάσταση ως απόλυτα χαόδη. Ε, Βεβαίω υπάρχουν προβλήματα, τα είδαμε και εμεί, αλλά και η Άννα και εγώ ο ίδιο και οι άλλοι συνάδελφοι ε, είμαστε συνηθισμένοι σε καταστάσει συγκρουσιακέ ή μετασυγκρουσιακέ και αυτό που είδαμε και αυτό που βρήκαμε στην. Λιβύη πόρο απέχει από αυτά που είχαμε δει παλιότερα στην Βοσνία, στο, στο Αφγανιστάν, σε ορισμένες χώρες της Αφρικής ε, μετά από τη σύραξη. Δηλαδή αυτό το χάος που περιγράφουν τα μέσα ενημέρωσης που κινδυνολογούν δεν ε, ε, είναι σωστό. Φυσικά η κατάσταση δεν είναι απλή, φυσικά τα πράγματα δεν είναι ε, αρμονικά και όμορφα, βεβαίως υπάρχουν ελλείψεις ε, όσον αφορά τις συμφωνίες, ε, κυρίως ο αφοπλισμός της Κατιμπά, της, μιλής, της αστυνομίας, αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί, προκύπτουν πολλές συγκρουσιακές καταστάσεις, διότι υπήρξε καταμερισμός των ζωνών που δεν λειτουργήσε καλά ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, προέκυψαν και ανοιχτές σειράξεις ε, μεταξύ των διαφόρων ομάδων και επομένως θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι να λειτουργήσει καλά ο στρατός, η αστυνομία, η στρατιωτική αστυνομία λειτουργούν ακόμα παραστατιωτικές οργανώσεις κτλ. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ευτυχώς δεν είχαμε γενικευμένες ε, σειράξεις και αντιπαραθέσεις. Επίσης ευελπιστούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ε, βοηθήσει τους Λίβιους που δεν ζητούν χρήματα ε, και αυτό είναι διαφορετικό από την αντιμετώπιση που είχαμε ε, σε άλλες σειράξεις όπου και σε άλλες προμηνικές καταστάσεις όπου η πρώτη μας κίνηση ήταν να οργανώσουμε ένα συνέδριο δωρητών και χορηγών. Στην περίπτωση της Λιβύης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ζητούν τεχνογνωσία, ζητούν πραγματογνώμα, ζητούν προσωπικό με γνώσεις έτσι ώστε να βοηθήσουν στον αφοπλισμό ε, και στην, ε, ε, στην σωστή επανεκκίνηση λειτουργίας του στρατού και της αστυνομίας. Υπάρχει ένα μεγάλο διοικητικό κενό το οποίο μπορεί να καλύψει με βοήθεια δική της Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναμειχθεί στο border management, διαχείριση των ε, συνόρων λοιπόν, γιατί είναι, ε, ε, είναι πάνω από 6.000 χιλιόμετρα τα σύνορα της Λιβύης, υφίστανται μεταναστευτικές ροές εξαιρετικά σημαντικές, γι' αυτό λοιπόν από την διάσκεψη των Παρισίων του Σεπτεμβρίου 2011 ήταν αυτό το θέμα της διαχείρισης των συνόρων ε, που ε, δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς οι διαδικασίες είναι ακόμα βαριές, είναι αργές, υπάρχουν ακόμα από πλευράς ε, Λιβύων κάποιες αργοπορίες, κάποια έλλειψη κατανόησης ενδεχομένως Έχουμε αυτή τη στιγμή μία αποστολή αξιολόγησης η οποία λαμβάνει η χώρα στη Λιβύη. Θα διαρκέσει δύο μήνες. Ε, θα έχουμε επίσης την δυνατότητα ε, να συζητήσουμε με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, το θέμα αυτής της αποστολής αξιολόγησης στη Λιβύη για να δούμε λίγο πώς έχει η κατάσταση. Ε, ήθελα να μοιραστώ κάποιες, κάποιες ε, εντυπώσεις ε, μαζί σας, γιατί για υπεριεντυπώσεων πρόκειται πέντε μέρες μείναμε επί τόπου. Ήταν πάρα πολύ βέβαια πυκνό το πρόγραμμα, εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να έχουμε μια γενική εντύπωση. Πρέπει να πω ότι εκτιμήσαμε ιδιαιτέρως ε, τους ε, συνομιλητές μας. Ε, είναι άνθρωποι ικανοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν με σαφήνεια, δεν ζητούν χρήματα, θέλουν να συνεχίσει η προσπάθεια που έδειξαν τα κράτη-μέλη στη διάρκεια της παρέμβασης στη Λιβύη και να συνεχίσει η βοήθεια αυτή με τρόπο σωστό, συντονισμένο και στοχευμένο. και ε, ε, βεβαίως ε, θα περιμένουν κάποια δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο. Γιατί ξέρετε καμιά φορά όταν μερικές χώρες αναλαμβάνουν δράσεις μόνες τους και η λιβική πλευρά δεν καταλαβαίνει ακριβώς περί τίνος πρόκειται και μπορεί να οδηγηθούμε και σε κάποιες παραφωνίες ή κάποιες κάποιες παρανοήσεις ο επικεφαλής ε, συνέλφος ε, Σαλαφράνκα ε, είναι αυτός ο οποίος ε, έστειλε την επιστολή στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως και ελπίζω ότι και στο μέλλον θα μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε το θέμα στην ΑΦΕΤ γιατί ξέρετε μπορεί τώρα και δικαίω οι προβολείς να έχουν στραφεί στη Συρία αλλά παρόλα αυτά η Λιβύη εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα εξακολουθεί να χρειάζεται την βοήθειά μας ε, η χώρα αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε και να δείχνουμε την προσοχή μας. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ ευχαριστούμε Άννα που θα μας παρουσιάσει στην γνωμοδότηση Α, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, κύριε Βανόρντεν, πριν, ναι, μπορούμε να... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα ε, την ε, αναφορά σας ε, στην επίσκεψη στη Λιβύη. Αναφερθήκατε και σε μια επιστολή τη στείλατε στα μέλη της Επιτροπής, γιατί διαφορετικά θα ήθελα να τη διαβάσω. Δεν την έχω διαβάσει ακόμα. Πρόκειται για ένα ζήτημα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα πρέπει να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Ε, έχοντας πλέον και από τη δική σας πλευρά ε, την γνώση του τι γίνεται επί τόπου. Θα ήθελα να διαβάσω και την επιστολή λοιπόν που εστάλει στην ε, Βαρόνη Άστον. Ναι, θα σας σταλεί η επιστολή, δεν έχει σταλεί ακόμα, θα σας σταλεί, τώρα διορθώνεται, είναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Ενδεχομένως το Προεδρείο της ΑΦΕΤ να έλαβε γνώση της επιστολής, αλλά βεβαίως ε, όταν είναι διαθέσιμη θα σας τη δώσουμε όσον αφορά για την εγγραφή στο σημείο, ε, σαν σημείο της ημερησίας διάταξης. Ναι, βεβαίως ε, θα ήταν και ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητούσαμε και με τον πρέσβη Hans-Georg Haber γιατί ακριβώς θα αναφερόμαστε στις πολιτικές δράσεις ε, της ε, κοινή πολιτικής ε, άμυνας ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει σχετικά με το τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει στο τραπέζι όσον αφορά τις μη στρατικές δράσεις κτλ. Αυτή τη βδομάδα, από όσον κατάλαβα, αύριο, αύριο και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα γίνει συζήτηση επί αυτού του θέματος. Θα ήθελα τώρα να συμπληρώσω κάτι μετά από αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος. Θέλω να σας εξηγήσω το εξής. Καλύτερα να τα πω αγγλικά. Πρέπει να σας πω ότι αυτές τις μέρες με εκλυπήσουν πάρα πολύ τα δημοσιεύματα του διότι ξέρουμε ότι ορτάζουν τις 17 Φεβρουαρίου, ένα χρόνο μετά την Επανάσταση. Και είμαστε εκεί και βλέπουμε ότι εμείς ε, με αγωνία τα αντιμετωπίζαμε το γεγονός, ότι φανταζόμαστε ότι θα υπήρχαν ε, κάποιες εκδηλώσεις και διότι κάποιοι πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ λεπτή και ασταθής ακόμη η κατάσταση. Δηλαδή, όλοι ενώθηκαν για να μπορέσουν να διώξουν αυτό το δικτάτορα, αλλά η διακυβέρνηση της χώρας αυτής δεν προοδεύει, δεν προχωρεί. Αυτό εν μέρει οφείλεται και στο θέμα της κατάστασης που αφορά την ασφάλεια. Και οι Ευρωπαίοι πιστεύουν βεβαίως ότι ε, αυτή η πολιτοφυλακή η οποία δημιουργήθηκε θα πρέπει να διαλυθεί. Πρέπει να πω όμως ότι είναι ε, τα μοναδικά άτομα αυτή τη στιγμή που μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια. Και δεν θα εξαφανιστεί εν μία νυχτή. Θα μείνουν για πολύ καιρό, διότι δεν υπάρχει στρατός. Δεν δουλεύει, αν θέλετε, δεν λειτουργεί ο στρατές, δεν λειτουργεί η αστυνομία. Άρα αυτή η πολιτοφυλακή είναι το μόνο όργανο, αν θέλετε, μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια. Και τα αιτήματα των Λιβύων από παντό είναι να τους βοηθήσουμε για την αποκατάσταση της ειρήνης και την αποκατάσταση της ασφάλειας. Όλοι αυτοί οι πολιταφύλακε δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται εδώ και καιρό. Όχι διότι δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει το διοικητικό πλαίσιο, αν θέλετε, για να διαθετήσει τέτοιου θέματα. Ζητούν λοιπόν από εμά και από γειτονικέ χώρες το ίδιο ακούμε, ότι η υποστήριξή μας είναι καλόδεχτη και απαραίτητη. Θα δείτε με, στην επιστολή που στείλαμε στη Lady Ashton. Actually call for Lady. Ζητούμε και από την ίδια την Lady Ashton και από όλου κάτι να κάνουμε από κοινού, στην πράξη. Να αφήσουμε τη ρητορική κατά μέρος. Αλλά πρέπει να ενεργήσουμε με πράξεις. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, αυτή τη στιγμή η βλέπουν ότι η παρούσα κυβέρνησή τους, η προσωρινή, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να γίνουν ε, ε, εκλογές, πρέπει να υπάρχει μια κάποια δομή. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να έχουν μια νόμιμη κυβέρνηση που θα παίρνει αποφάσεις. Δεν πρέπει να περιμένουν να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, πρέπει αμέσως να τους βοηθήσουμε και με κάποια μέτρα που θα εξασφαλίσουν ε, όχι μόνο κάποιες ε, δικές μας αποστολές, αλλά τη μόνιμη παρουσία μας και με πιο δομημένο τρόπο να βοηθήσουμε ε, την αποκατάσταση της κοινωνίας, τον αφοπλισμό, της δεδομένου ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά και είναι θέμα ασφάλειας γενικότερα και δική μας ασφάλειας. Εδώ δεν διακυβεύεται μόνο η ασφάλεια της ε, Λιβύης. Δεν υπάρχει μόνο το θέμα του εξισουσίας που πέρασε από τα χέρια του Καντάφη σε αυτούς τους επαναστάτες. Είναι θέμα ασφάλειας γενικότερο. Δεν υπάρχουν έλεγχοι πουθενά είναι διαπερατά τα σύνορα, η γενικότερη ε, περιοχή λοιπόν έχει πρόβλημα ασφάλισης. Θα, θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα το θέμα αυτό. Τώρα, πριν να ξαναδώσω το λόγο στην Άννα τώρα, λέει ο Πρόεδρος, για να συζητήσουμε για την ε, εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική της. Για την έκθεση αυτή τι οποίε συντάξει αγνομοδότησης είναι οι αναγκόμενε. Γκόμε έχουμε 42 τροπολογίες και η ψηφοφορία τη έκθεση θα γίνει στην ΑΦΕΤ την πέμπτη το πρωί. Άννα λοιπόν, έχει το λόγο και μετά θα δώσουμε το λόγο στους κοιόδες συζητητές. Έχω συντάξει την ε, ε, γνωμοδότησή μου και έχω και εγώ καταθέσει κάποιες τροπολογίες στην εκθεσή μου, διότι είχα πάρα πολύ λίγο χρόνο για να παρουσιάσω την αρχική μου νομοδότηση και μετά όταν είχα περισσότερο χρόνο ξαναείδα το κείμενό μου και προσπάθησα να ενεργήσω με πρακτικό πνεύμα. Νομίζω ότι η προστιθέμενη αξία της ΦΕΤ και των απόψεων της δικής μας Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε from uh, I mean, uh, from the, the narrow perspective of από την στενή προοπτική της εσωτερικής ασφαλείας για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να επιλύσουμε και θέματα που από της εξωτερικής στρατηγικής ασφάλειάς μας. Πρώτα απ' όλα, διότι κάποιες απειλές είναι ταυτόσιμες και κάποιες από τις οποίες δεν μπορούν να επιληθούν με μέσα τα οποία είναι αποκλειστικά ή εσωτερικού ευρωπαϊκού χαρακτήρα ή εξωτερικού. Υπάρχουν ο διασυνοριακός, ο παγκόσμιος χαρακτήρας των προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια. Άρα πρέπει να έχουμε μέσα κοινά για να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο επικοδομητική γίνεται, μιλώντας κυρίως για θέματα που αφορούν την ασφάλεια, δεδομένου ότι τώρα διαθέτουμε και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εσωτερικής Δράσης και χρειαζόμαστε πολύ καλύτερο ε, συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών της κυρίας Άστον, ε, του, του, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και όλων των άλλων ε, σχετικών θεσμών που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα προσπάθησα να τα εξηγήσω στην εκθεσή μου και στις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σε θέματα στρατηγικής για την ασφάλειά μας εσωτερική και εξωτερική, που θα πρέπει να βασίζεται πρώτα απ' όλα στην προσέγγιση της ασφάλειας των ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό συνάδει ούτως ή άλλως και με τον θεμελιώδη στόχο μας, που είναι ε, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτος δικαίου, σεβασμός της δημοκρατίας σε εσωτερικό και σε έξω κοινοτικό επίπεδο. Όπως επίσης ανέφερα, λέω πόσο σημαντικές είναι και οι διάφορες ε, αποστολές ε, οι οποίες αναλαμβάνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν και την εσωτερική και την εξωτερική μας ε, ασφάλεια. Σκέφτομαι την τρομοκρατία. Σκέφτομαι σχέσεις που μπορούσαμε να αναπτύξουμε με τις γειτονικέ χώρες μας ε, νοτίως της Μεσογείου μετά από τις εξελίξεις του τελευταίου χρόνου την Αίγυπτο και σε άλλες χώρες και νομίζω ότι είναι γελίο να παραγνωρίσουμε κάποια μέσα που μας παρέχονται, που είναι στη διάθεσή μας και θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της αντιμετώπισης της εσωτερικής ασφάλειας. so far in a Υπάρχει ένα άλλο τομέα στον οποίο έχουμε κενά και θα πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα. Είναι ο τομέας του ειδικού συντονιστή για θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της διασύνδεσης των προσπαθειών με αυτές που καταβάλλονται από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Εσωτερικής Δράσης που δημιουργήθηκε σαν ε, ένα μέσον προάσπισης της ασφάλειας. Πολλές φορές το τι έχει γίνει σε αυτό το τομέα από μας παραγνωρίζεται και θα πρέπει, όπως λέγω, να συντονιστούμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο. Ο Μάικλ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Πρέπει να πω ότι εμείς στο ΕΛΚ βασικά συμφωνούμε με την έκθεσή σας, έχουμε βεβαίως να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις και μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Γιαννάκου που είναι η σκιώδη μας, η οποία δεν μπορεί σήμερα να παρευρεθεί στην συνεδρίασή μας, διότι αυτή τη στιγμή είχε πάει στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρέμεινε και η κυρία Γιαννάκο, όπως και άλλοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την καταπολέμηση τρομοκρατίας. Πιστεύουμε ότι δεν είναι ε, αρκετά όριμη η ιδέα που εκφράζεται για τις ε, ομάδες εργασίας τις οποίες αναφέρεστε εσείς για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους θεμάτων. Πρέπει να πω ότι προς το παρόν μόνο τρία άτομα ασχολούνται με αυτά τα θέματα και δεν υπάρχει ακόμη ε, ε, ο κατάλληλος εξοπλισμός και να μεταφέρουμε εκεί τις, κάποιες αρμοδιότητες ίσως είναι πολύ ενωρίς. Όταν θα έχουμε εκεί τον κατάλληλο εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό, ίσως να είναι σωστή η πρότασή σας. Θα έπρεπε ίσως να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση θα πρέπει να βασιστεί περισσότερο στην ε, πραγματογνωσύνη της ε, αντιτρομοκρατικής. Στην παρούσα πραγμάτα, κατάσταση λοιπόν των πραγμάτων είμαστε κατά της τροπολογίας αυτής, όχι για θέματα αρχής, αλλά διότι η πραγματική κατάσταση είναι διαφορετική. Δηλαδή ε, δεν έχουμε τις απαραίτητε, τους απαραίτητους πόρους. Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία, τη συμβαστική τροπολογία 4. Ένα μέρος της φράσης χάθηκε εδώ. Εκεί που γίνεται λόγος για τις αποστολές που αφορούν την ε, κοινή ασφάλεια, άρα ε, είμαστε κατά της ε, συμβαστικής τροπολογίας 4. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι για μεγάλη ευχαρίστηση είμαι σήμερα εδώ. Διότι ως τακτικό μέλος πάντα θα πρέπει να είμαι παρόν συνεδριάς υπό Επιτροπή Ασφαλείας Άμυνας. Σπάνια όμως το κάνω, διότι παρόλο ότι την αγαπώ αυτή την Επιτροπή, συμπίπτει πάντα με τις εργασίες κάποιες άλλες. Λοιπόν, σήμερα χαίρομαι που μπόρεσα να είμαι εδώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Άννα Γκόμες, διότι εδώ και χρόνια βλέπω πώς έχει αναλάβει την μελέτη του θέματος αυτούς και σιγά σιγά μαζεύει τα κομματάκια του πάζελ που λέγεται κοινή ασφάλεια εσωτερική και εξωτερική. Όταν στο παρελθόν είχε προταθεί μία πρόταση ε, πρωτοβουλίας για την εξωτερική διάσταση της ασφάλειας στα πλαίσια της διεθνούς τρομοκρατίας Είχα κάνει εγώ την έκθεση με δική της πρωτοβουλία. Λοιπόν, ότι και τώρα και πάλι στο πάζελ αυτό προσθέτουμε ένα νέο κομματάκι. Συμφωνώ με το περιεχόμενο της ε, έκθεσής της και με τις ε, συμβαστικές της τροπολογίες. Απλώς θα ήθελα, όχι για να αναπτύξω εδώ μια νέα έννοια η οποία μας απασχολεί, σε απασχολεί πάρα πολύ στην Ισπανία, θα έχετε ακούσει να γίνεται λόγος για την τριπλή διαδικασία η οποία έχει αναλυφθεί κατά του δικαστή Γκαρθών. Όπως ξέρετε, έχει ασχοληθεί με τη διαφθορά και στα πλαίσια μεταξύ άλλων αυτού του θέματος ασχολήθηκε και με την υπόθεση Γκούρτελ και για να μπορέσει να επιλύσει το θέμα αυτό, ε, ακολούθησε την, ε, οδηγήθηκε σε παρακολούθηση κάποιων τηλεφωνημάτων μεταξύ των υπόπτων, όχι για άλλο λόγο, αλλά για να μπορέσει να μαζέψει στοιχεία και να πολεμήσει το θέμα αυτό. Το ε, δικαστήριο απεφάνθη ότι αυτό δεν ήταν σωστό στη δικασία, τον καταδίκασε. Το θέμα τώρα εδώ δεν είναι να υπερασπιστούμε τον δικαστή Γαρθών που ξέρει και το κάνει αυτό εξαιρετικά μόνος του. Αλλά θα ήθελα εδώ να εκφράσω μια μεγάλη ανησυχία διότι κανένας δικηγόρος δεν μπορεί ακόμη σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν το επιτρέπει ο νόμος δεν μπορεί να παρακολουθεί ένα τηλέφωνο διότι κινδυνεύει να τον καταδικάσουν οι συνάδελφοί του. Όπως στην περίπτωση του Γκαρθών. Καταδικάστε λοιπόν για κάτι για το οποίο δεν έχει καταδικαστεί κανένας από το μεγαλύτερο στην ε, ιστορία αυτού του δικτύου διαφοράς Γκούρτελ να έχει καταδικαστεί. Κανένας από αυτούς δεν καταδικάστηκε. Και κανένας δεν έχει κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ό,τι γίνει θα δημιουργήσει ε, προηγούμενο και στην Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να διαταράξουμε την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ του πόσο αποτελεσματικοί πρέπει να είμαστε για να καταπολεμήσουμε την τροπολογία και συγχρόνως πώς πρέπει ε, να εγγυόμεθα τα δικαιώματα υπεράσπισης ακόμη και των κατηγορημένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι οι τροπολογίες που εσείς οι ίδιοι υποβάλλετε στην έκθεσή σας, στην, ε, ε, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ το κείμενο. Έχω υποβάλει τροπολογίες κι εγώ. Μία φορά τους μηχανισμούς συντονισμού ανάμεσα στην Υπηρεσία εξωτερική... Εξωτερικών Δράσεων ε, και την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων. Δεν είμαι ε, σίγουρη ότι υπάρχει τέτοια συνεργασία ε, και λέμε να την εντείνουμε. Θα μπορούσα να πούμε να την βελτιώσουμε. Αλλά λέω απλώς ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο, να την ενδυναμώσουμε. Επίσης, ε, Ε, αυτά τα situation centers ε, νομίζω ότι έχω υποβάλει μια τροπολογία γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί ε, για να, και να περιμένουμε λίγο τις θεσμικές διαδικασίες πιο προσεκτικοί να είμαστε. Και υπάρχει και άλλη μία τροπολογία, ίσως επί της ουσίας να είναι και πιο σοβαρή. Αφορά την ε, παράγραφο που λέει ότι θα πρέπει ε, να λαμβάνονται υπόψη ε, σωστά οι κίνδυνοι οι απειλές μάλλον, τρομοκρατικές απειλές και να οργανώνονται από κοινού οι δράσεις, η καταπολέμηση αυτών των απειλών κτλ. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι ε, είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσει κανείς ε, στρατιωτικές δυνάμεις ε, για αντιμετώπιση εσωτερικών προβλημάτων ασφάλειας. Και επομένως, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον σύμφωνα και με το γερμανικό σύνταγμα, μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Ξέρω ότι οι παραδόσεις διαφέρουν στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά για μας είναι δύσκολο λαμβάνοντας υπόψη και την γερμανική ιστορία και το παρελθόν, έχουμε πρόβλημα με αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί. Ε, είδατε τις τροπολογίες μας, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο ε, και πιστεύω ότι θα βρούμε και συμβιβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόεδρος, άλλοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν παρατηρήσεις. Άννα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, για τα σχόλια και τη συμβολή τους ε, στο θέμα αυτό. Έχω υποβάλει μεταξύ και προφορικές, συγγνώμη, συμβιβαστικές τροπολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των διαφόρων συναδέλφων όσον αφορά αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κάποιο συμβασμό με τον Μάικ Γκάλλαρ και τους ε, συναδέλφους από τη δικιά του ομάδα ε, όσον αφορά ε, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και την ομάδα εργασίας. Ναι, αλλά η ίδια η ουσία είναι εκεί. Δηλαδή θέλουμε μια ομάδα η οποία θα ασχολείται με την εξωτερική όψη των τρομοκρατικών απειλών. Ενδεχομένως μπορούμε να βρούμε κάποια άλλη διατύπωση, κάποια ε, λύση που να μας ε, ευχαριστεί όλους και που θα προετοιμάζει κατά κάποιο τρόπο το έδαφος για μια καλύτερη εξέλιξη. Ε, δεν έχω ε, αφήσει, δεν έχω ξεχάσει την αναφορά στην ε, κίνητη πολιτικής ασφάλειας ε, και άμυνας. Το, έβαλα την αναφορά, την έβαλα κάπου αλλού. Κάπου είναι τώρα, δεν, δεν την βρίσκω αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρω ότι η αναφορά στην ΚΠΑ υπάρχει. Η ΚΠΑ δεν είναι, αφορά απλώς και μόνο στρατιωτικές αποστολές. Υπάρχουν και άλλες αποστολές. Η ε, Γιούλεξ ε, στο Κωσυφοπαίδιο ε, βεβαίως δεν είναι στρατιωτική, είναι πολιτική. Είναι μη στρατιωτική. Και επομένως οι φόβοι της Φρανσέσκα δεν επαληθεύονται εδώ. Θέλω να πω ότι Μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν ε, τέτοιες ε, ε, τέτοιε διαδικασίες. Δηλαδή και οι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει η αποστολή Γιούλεξ στο Κωσυφοπαίδιο ενδεχομένως ε, να μας ενδιαφέρουν ε, και μετά από σωστή επεξεργασία αυτές οι πληροφορίες της Γιούλεξ θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στο ένα ή στο άλλο πράγμα και επομένως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τέτοιες πληροφορίες για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά τότε θα πρέπει να το γράψετε ότι είναι μη στρατιωτικές αποστολές της ε, ΚΠΑ. Φανταστείτε ότι έχουμε μια κοινή πολιτική και στρατιωτική αποστολή στο μέλλον στη Λιβύη της ε, ΚΟΥΠΑ. ΚΠΑ. Ε, μπορεί να γίνει αυτό, δεν λέω ότι θα γίνει αύριο, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο του μέλλοντος. Και αυτή η αποστολή, ας πούμε, θα εκπαιδεύει το στρατιωτικού, θα εκπαιδεύει το στρατό, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά θα ασχολείται και με άλλα θέματα, εκτός από αυτά τα οποία είναι μη, μη στρατιωτικά. Εκπαίδευση αστυνομικών κλπ. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή η αποστολή ε, έχει βρει, έχει ε, αναγνωρίσει έναν κίνδυνο στη Λιβύη Ε, ο οποίος κίνδυνος αυτός μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε εμάς. Τι θα κάνουμε, θα αγνοήσουμε αυτή την προειδοποίηση περί ενδεχομένου κινδύνου επειδή προέρχεται από στατιωτική πηγή. Δεν νομίζω το θέμα είναι αυτές τις πληροφορίες. Θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, σωστά. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Έτσι ώστε να γίνουν σεβαστές οι θεμελιώδεις ε, ε, προϋποθέσεις, οι του νόμου, το διεθνές δίκαιο κλπ. κλπ, κλπ. Υπό τους όρους αυτούς μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Όσον αφορά τώρα ε, τις επιφυλάξεις ε, για τους πολίτες. Ε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όμως προέρχομαι από μία χώρα όπου η αστυνομία ήταν λίγα αποτελεσματική και δεν τη συμπαθούσαν και πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ σημαντική η υπηρεσία αυτή για την ΙΣΙΤΣΕΝ είναι μία ε, οργάνωση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για την ανάλυση, την αναλυτική διαδικασία framework in this articulation between the tools that we use for addressing the internal Λοιπόν, γιατί να μην εμπλακεί και η Citizen, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσουμε, ιδίω ε, αν υπάρχει ο κίνδυνος από εξωτερικές πηγές. Γιατί να περιοριστούμε, γιατί να αποκοπούμε από αυτό το εργαλείο, από αυτό το μέσον το οποίο υπάρχει διατίθεται και το οποίο μέσων αυτών, η Citizen δηλαδή, θα πρέπει να σέβεται ορισμένους κανόνες οι οποίοι είναι σαφώς προδιαγραμμένοι. Γι' αυτό δεν συμμερίζουμε τις επιφυλάξεις και τις φοβίες που εκφράζουν ορισμένοι συνάδελφοι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε την οργάνωση αυτή, αυτό το, το φορέα αυτών που διατίθεται, που είναι στη διάθεσή μας. Ο τρόπος είναι πολύ σημαντικός. Μπορούμε να έχουμε μεγάλο όφελος από την ε, συνεργασία μαζί τους. Ο Πρόεδρος. Για το θέμα αυτό που απασχολεί την Φραντζίσκα περισσότερο. Υπάρχει διερμηνία στα γερμανικά, βεβαίως. καλύτερα να εκφραστώ στα γερμανικά, διότι άπτεται τη εσωτερική ασφάλεια, που στη Γερμανία είναι εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Η εσωτερική ασφάλεια ε, και ο παραλληλισμός ή αν θέλετε η ισοτιμία με την στρατιωτική ασφάλεια ε, δημιουργεί αντιδράσεις και γι' αυτό θα έλεγα να περιστούμε στην, να διατυπώσουμε αποστολές της ε, ΚΠΑ και να αφήσουμε όλα τα άλλα. Διότι υπάρχουν διαφορετικές ιστορικές πολιτιστικές προσεγγίσεις και απόψεις. Όταν μπλέκονται οι στρατιωτικές και μη στρατιωτικές πτυχές, ε, εάν είναι civilian, δηλαδή πολιτικές μη στρατιωτικές αποστολές και αν ούτως ερμηνεύσουμε ε, το περιεχόμενο τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή να διευκρινίσουμε όπως είπε και η Άννα όταν πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει, δεν τίθεται πρόβλημα να πλουστεύσουμε τα πράγματα και όχι να τα περιπλέξουμε. Ο κ. Γκάλερ. Ευχαριστώ. για μας. Ε, η συνάδελφος αυτή μιλάει εκ μέρους των πρασίνων. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι καλύπτει όλους. Εγώ συμφωνώ με την Άννα περισσότερο. Ε, υπάρχουν αρνητικές εμπειρίες ε, από το παρελθόν, ε, από ιστορικής πλευράς και γι' αυτό πολλές φορές στο παρελθόν ζητούσαμε μια αυστηρή διαφοροποίηση, έναν αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σκέλους. Όμως η συγήτρια ε, βασίζεται στο γεγονό ότι τώρα οι δημοκρατικοί θεσμοί έχουν προχωρήσει τόσο ώστε να μην χρειάζεται πλέον αυτή η απομόνωση, αυτός ο αυστηρότατος διαχωρισμός και να υπάρχει μία συνέργεια μεταξύ των δύο σκελών. Γι' αυτό πιστεύω ότι μία τέτοια ειδική ε, συζήτηση ε, ε, που άπτεται του εθνικού επίπεδου δεν θα ήθελα να τη δω να μεταφέρεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ συμφωνώ με την εισηγήτρια, με την Άννα Γκόμες και... Πολύ καλά. Ετοιμιγωρία την Πέμπτη το πρωί. Δεδομένου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την 1η Μαρτίου η έκθεση αυτή. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ο κύριος πρέσβης Χάμπερ ζήτησε συγγνώμη. Θα έχουμε την ευχαρίστηση να τον δούμε κάποια άλλη φορά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τις μη στρατιωτικές αποστολές. Ευχαριστώ.